Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τη δήλωση της ΥΠΑ της εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας μετά από τη συνάντηση κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας της 31ης Μαΐου και 1ης Ιουνίου. Το λόγο έχει η Αντιπρόεδρος κυρία Άστον. Uh, κυρία Πρόεδρε, Αξιότιμα μέλη, χαίρομαι που έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να συζητήσουμε το αποτέλεσμα της τελευταίας διάσκεψης κορυφής Ευρωπής ε, Ρωσίας, το Ρώστοφετον. Ήταν πάρα πολύ καλή συνεργασία, επικοδομητική και επιβέωση την ε, επιθυμία της Ρωσίας για πιο στενέ σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη διάσκεψη της αυτή ξεκινήσαμε την εταιρική σχέση για εξυγχρονισμό. Όπως πολλοί από τους ε, βουλευτές γνωρίζουν, ο πρόεδρος Μοντεβέλες λέει συνεχώ ότι θα πρέπει να εξονιστεί η Ρωσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν ο μεγαλύτερος ε, εμπορικό εταίρο τη Ρωσία ε, συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος ότι για είναι επιτυχής οποιαδήποτε προσπάθεια εξοργανισμού θα πρέπει να είναι ευρεία, να καλύπτει επιχειρησιακό πνεύμα, καινοτομία και να ενδυματωμώσει τις δημοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου. Θα πρέπει η κοινωνία των πολιτών να συμμετάσχει σε κύριους τομείς του εξυγχρονισμού. Ε, Επίση, ε, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά του προασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι πρόσθετε διαδηλώσει ε, είναι απόδειξη των προβλημάτων που υπάρχουν. Επίσης, η αστάθεια στον Κάφκασο είναι άλλος τομέας προβληματικός. Υπήρξαν όμως και θετικές εξελίξεις που πρέπει να τις αναγνωρίσουμε. Η διεύρυνση του μορατόριου για τη θανατική ποινή και η έγκριση του πρωτοκόλλου 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το κράτο δικαίου και η καταπολέμηση τη διαφθοράς θα οδηγήσουν σε πιο φιλική προς επιχειρήσει περιβάλλον, φιλικό περιβάλλον. Η Ρωσία καταλαβαίνει ότι θα πρέπει να κάνει περισσότερα για να προσελκύσει επενδυτέ, Το ενταχθεί στο Παγκόσμιο Οργάνωση Εμπορίου είναι ένα δείγμα του το θα μπορούσε να γίνει και ελπίζουμε ότι θα μπορούσε να ολοκληρώσουν τις σχετικές εργασίες για την ένταση στην ΠΟΕ. Η πολιτικές δηλώσεις θα πρέπει να μεταφραστούν σε πραγματικότητα. Η εφαρμογή της ε, Τελωνιακής Ένωσης Ρωσίας-Καζακστάν ε, δεν έχουμε μας κανένα πρόβλημα με αυτές τις τελωνιακές ενώσεις. Ε, είμαστε μια τελωνική ένωση, αλλά αυτή που προτείνεται στη Ρωσία παρεμποδίζει το εμπόριο, δεν το ευνοεί και αυτό δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Επίση, θα πρέπει να υπάρχει μια νομική βάση για τι σχέσει στον τομέα τη ενέργεια. Ο εκνευρισμό τη πολιτική θα παίξει σημαντικό ρόλο. Θα πρέπει να υπάρχουν σημαντικέ διατάξει στη Νέα Συμφωνία που θα αντικατοπτρίζουν τι αρχέ ε, τη συνθήκη για την ενέργεια. Επίση, ελπίζουμε ότι η χάρτα αυτή για την ενέργεια θα, θα καταστεί ένα βήμα για να συζητηθούν πολλά άλλα σχετικά θέματα όπω υποδομέ. Εμείς ενθαρρύνουμε τη Ρωσία να είναι πιο φιλόδοξη στους στόχους της που τώρα είναι 15 έως 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για τη μείωση του δοξιδίου του άνθρακα. Η Ρωσία καταλαβαίνει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το ευαίσθητο θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, συμφωνεί η Ρωσία να προχωρήσει βήμα προς βήμα. Υποβάλαμε συγκεκριμένες προτάσεις Επίσης όσον αφορά τη διευκόλυνση της θεώρησης των διαβατηρίων. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε σύντομα να δούμε να έχει ολοκλήρωση η προσπάθεια για διευκόλυνση των διέλευτων συνόρων για τους Πολωνούς και τους Ουκρανούς, πράγμα που θα διευκολύνσει αυτούς που ζουν στο Καλίνιγκραντ. Επίσης, θέλουμε να δούμε κατά πόσο μπορούμε να εξελίξουμε περαιτέρω τη συνεργασία τύπου Αταλάντη. Προφανώ η αυτονομία για τη λήψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να παραμείνει ω έχει. Στη διάσκεψη κορυφή συζητήσαμε επίσης και διάφορα διεθνή θέματα όπως το ε, πυρηνικό πρόβλημα του Ιράν, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, το Κόσοβο ε, και χαίρηκα για την κοινή δήλωση που έκανε ο Πρωθυπουργός Λάροφ και εγώ για την απώλεια ζώων κατά τη διάρκεια του επεισοδίου αυτού στη Γάζα. του λεχθέντος, οι άποψεις μας διαφέρουν όσον αφορά το κοσυγοπαίδιο, τη Μολδαβία, όπου δεν υπάρχει η σωστή ρωσική στάση. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στους ομιλητέ από τι πολιτικέ ομάδε. Θα αρχίσουμε από το ΑΕΛΚ για δύο λεπτά. Ο κύριο Μπρόκ. Είπατε εκπρόσωπε, αντιπρόεδρε τη Κομισιόν, κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω κυρία Άστον για την παρουσίασή σα και τον τρόπο με τον οποίο οργανώσετε τη διάσκεψη κορυφή. Είναι σαφέ νομίζω ότι υπάρχουν ανησυχίε ότι ορισμένε, όσον αφορά ορισμένε εξελίξεις κράτους δικαίου στην Ρωσία, όσον αφορά τις διαδηλώσεις όσον αφορά την γεωργία που δεν υπάρχει το δίκαιο των εθνών, δεν ισχύει. Από την άλλη μεριά ότι υπάρχει και κάποια πρόοδος, όπως παραδείγματος χάρη συμφωνία για τον εξορισμό που θα συμβάλλει σημαντικά για να προχωρήσουμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ρωσία έχει για μας μεγάλη στρατηγική σημασία. Έχουμε μεγάλα κοινά συμφέροντα στον οικονομικό τομέα, στον ενεργειακό τομέα και είναι σαφές νομίζω ότι οι διαπραγματεύσεις 5 είναι 1 για το Ιράν και το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών καταλήξαμε σε μια κοινή θέση. Αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό. Όπω και για άλλα θέματα, η ενδυνάμωση παραδείγματο τη εργασία του κουαρτέτου για τη Μέση Ανατολή είναι επίση μεγάλη σημασία και θα πρέπει να προχωρήσει. Από την άλλη μεριά είναι και θέμα αξιοπιστία τη Ρωσία, Ο τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τη νέα συνθήκη ε, εταιρική σχέση και σχέση γυπνίασης σε διάφορα θέματα, όπως παραδείγματο χάρη το τεράστιο θέμα της ενέργειας που μέχρι στιγμής διακανονίζεται στην ενεργειακή κάρτα και δεν εφαρμόζεται. Η Ρωσία θα πρέπει να είναι έτοιμη να δεσμεύεται οικονομικά για τις συμφωνίες αυτές. Όπως παραδείγματο χάρη θα πρέπει να είναι έτοιμη να λάβει σοβαρά υπόψη τις διαπραγματεύσεις ΠΟΕ και να γίνει πλήρως μέλος σε αυτό το διεθνέ βήμα άρα θα πρέπει να δεχθεί και η ε, Τελωνική Ένωση με το Καζαχστάν και τη Λευκορωσία να κατανοήσει ότι δεν είναι το καλό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρόκειται για θέμα ε, αξιοπιστίας σχετικά και με τις δεσμεύσεις για την ομάδα του G20. Το θέμα της θεώρησης των διαβατηρίων θα πρέπει επίσης να προωθηθεί, αλλά δεν θα πρέπει αυτό το θέμα να συσχετιστεί με τις θεωρίες των ε, ε, διαβατηρίων των ανατολικών μας γειτόνων, γιατί δεν επιτρέπεται από την Ουκρανία να μπορεί κανένα να έρθει πιο εύκολα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα ρωσικό διαβατήριο από ότι με ένα ουκρανικό. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος των σοσιαλιστών και δημοκρατών, ο κύριος Σεβερίν, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Ήπατη εκπρόσωπος, αγαπητοί συνάδελφοι. Οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσία έχουν μεγάλη στρατηγική σημασία. Χαρακτηρίζονται όχι μόνο από τα οικονομικά μας συμφέροντα και από το στόχο της στενής συνεργασίας σε πολλούς διεθνούς, διεθνείς τομείς. Από γεωγραφική άποψη η Ρωσία είναι και θα παραμείνει ο πιο κοντινός γείτονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εξακολουθεί να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρωασιατική αλλά και στην, στον ευρωασιατικό αλλά και στον ευρωατλαντικό χώρο. Υπάρχει συμπληρωματικότητα μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία σε ό,τι αφορά τι ανάγκε, του πόρου και τη σύμπτωση, τη σύγκληση ορισμένων στόχων παγκόσμια σημασία. Πρέπει να αντιληφθεί κανεί ότι μια σταθής ευάλωτη και προβληματική στο εσωτερικό της Ρωσία ε, θα είναι μια πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αντίθετο αποτελεί σταθερότητα. Είναι καλύτερο λοιπόν παράλληλα να έχει κανείς ένα σταθερό και όχι έναν ευάλωτο και ασταθή γείτονα. Οι στρατηγικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσία πρέπει να ενισχυθούν σε πολλούς τομείς. Σύμπραξη για εξυγχρονισμό, κάτι το πολύ σημαντικό που θα συμβάλλει στη δημιουργία εμπιστοσύνης, και σύγκλησης με τη Ρωσία σε βρεις τομεί κοινού ενδιαφέροντος. Εταιρική, έσχυση, σχέση, σύμπραξη για προσχώρηση στον ΠΟΕ πρέπει επίσης να εξεταστεί και θα διευκολυνθεί, θα διευκολυνθεί η Ρωσία για την ένταξή της με την υποστήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει επίσης να ενισχυθεί μια τριμερής συνεργασία με τις χώρες υπομετάβαση. μετάβαση πρέπει να σκεφτούμε μια τριμερή σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείε επίσης για την ενίσχυση και την μεταρρύθμιση των διεθνών, των παγκόσμιων ρυθμίσεων σε ό,τι αφορά την ε, ειρήνη και την ασφάλεια πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε το θέμα των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων με σωστό τρόπο να μην το θεωρήσουμε σαν εργαλείο γεωστρατηγικό, αλλά σαν ε, το θεμέλιο μιας πραγματικής συνεργασίας σε όλους τους τομείς. Ευχαριστώ για την άλλη ο κύριος Όγιουλαντ. Η κυρία Όγιουλαντ, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Η η διάσκεψη Ρωσία Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ροστοβαντών μας γέννησε με ελπίδες σε ό,τι αφορά ειδικό την οικονομική συνεργασία, αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε τις αρχές της δημοκρατίας, των ανθρώπινων και πολιτικών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου καθώς αναπτύσσεται η συνεργασία μας το πρόγραμμα εξυγχρονισμού έχει σκοπό να διαφοροποιήσει το οικονομικό περιβάλλον και να προωθήσει τι εμπορικέ σχέσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο μπορεί να επιτευχθεί σε περίπτωση που λάβει όλα τα μέτρα η Ρωσία για να βάλει τάξη στο δικό τη χώρο, στο δικό τη περιβάλλον. Η Τελωνική Ένωση Ρωσία, Καζακστάν και Λευκορωσία μα δείχνει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να προσχωρήσει άμεσα στον ΠΟΕ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αποτέλεσμα να απομακρύνονται ε, ε, δυνητικοί ε, επενδυτές από τη Ρωσία. Θέλουμε μεγαλύτερη ασφάλεια στον τομέα της ενέργειας και σε όλους τους άλλους τομείς. Θέλουμε μεγαλύτερη προθυμία από πλευρά της Ρωσίας για ευρύτερη συνεργασία σε διακινήσεις αγαθών και πρέπει επίσης να απλοποιηθεί το σύστημα των θεωρήσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Πρέπει λοιπόν να λάβει πρακτικά μέτρα η Ρωσία για την ενεργειακή ασφάλεια. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσει με τη Ρωσία και να υπογραφεί μια συμφωνία που θα στηρίζει την αρχεία της ε, ενεργειακής ασφάλειας ε, θέλουμε να επικυρώσει το πρωτόκολλο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης ανθρώπινα δικαιώματα η Ρωσία και επιβεβαίωση του δικαιοστασίου για την θανατική ποινή. Θέλουμε παράλληλα να τονίσουμε ότι πρέπει να κληρώσει υποχρεώσει η Ρωσία απέναντι στη Γεωργία και προσβλέπουμε στην ειλικρινή συνεργασία της για την επίλυση των διαφορών στο Νότο Κάφκασο και τη Μολδαβία. Θέλω να υπογραμμίσω κάποιες σημαντικές εξίε που πρέπει να χαρακτηρίζουν τη σχέση μας με τη Ρωσία σε όλους τους τομείς. Δεν μπορούμε να δεχθούμε παραβιάσεις των ανθρωπών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Κανένα οικονομικό όφελος δεν μπορεί να είναι πιο σημαντικό από τις αξίες που εκπροσωπεί ε, και εκφράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δεύτερη δίκη του Μιχαήλ Χοντακόφσκι είναι ένα παράδειγμα μη τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου από τη Ρωσία. Η τροπολογία 5 το τονίζει αυτό και καλούμε για αυτό τους συναδέλφους να την υποστηρίξουν. Για την ομάδα των Πρασίνων, ο κύριος Σούλτς για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, έχουμε μπροστά μας ένα ψήφισμα για το αποτέλεσμα της Έσχεσης Κορυφής Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλες τις προσπάθειες του Πρόεδρου Μέρκεφ να εξυγχρονίσει, θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι ο εξυγχρονισμός δεν είναι μόνο τεχνικό θέμα. Πολύ την κατάνοση που η Ρωσία θέλει να αναπτύξει την νανοτεχνολογία και να αναπτύξει μια κοιλάδα σιλικόνης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι χρειάζεται και μια κοινωνία των πολιτών ζωντανή, στην οποία μπορούν να αναπτυχθούν οι καινοτομικέ ε, ε, τάσεις. Μια τέτοια εταιρική σχέση θα πρέπει να προσφέρουμε στη Ρωσία και γι' αυτό θα πρέπει να ξεπεράσουμε τα ελλείμματα και να αναφερθούμε στα προβλήματα όπως έκανε ο πρόεδρος Φαν στο Ρόστοφ και η κυρία Άστον εδώ. Θα πρέπει αυτά όμως να αντικατοπτρίζονται και στο δικό μας ψήφισμα και γι' αυτό υποβάλαμε ε, τέσσερις τροπολογίες που σας παρακαλούμε να υποστηρίξετε. Πρόκειται για τη λήξη της πολιτικής δίωξης, βελτίωση στην ποινική δίωξη, την άρση του στρατηγικής ποινής του Αντρέη Σαββόσκη και την απελευθέρωση του κ. Πασοκόψη και Λεμπεντιέφ, τέλος των ανθρωπιστών στο Κάφκασο και την ελευθερία του συνέρχεστε που εγγυάται και το Ρωσικό Σύνταγμα. Η εξωτερική ελευθερία θα πρέπει δηλαδή να σχετίζεται άμεσα με την εσωτερική ελευθερία, γιατί πιστεύουμε και η Ρωσία δεν μπορεί να είναι διαιρετή η ελευθερία. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Τάνοκ για, το συνταγμα... για την ομάδα του για ένα λεπτό. Πρόεδρε, λέει Άστον, ε, βλέποντας ε, ε, το πλησίον της Ρωσίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οικονομία σας τριών εκατομμυρίων και τα αποθέματα ε, αερίου που έχει, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική χώρα, ιδίω και μέσα στα πλαίσια του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και της κατάστασης στη Βόρειο ε, Κορέα και στην ε, Μέση Ανατολή και όσον αφορά τα πυρηνικά όπλα του Ιράκ και το να πιέσει την Τουρκία να ανοίξει τα με την Αλμονία. Έχουν βελτιωθεί οι σχέσεις βέβαια μεταξύ Μόσχας και Κίεβου, αλλά το να επιτραπεί στη Ρωσία να μπορέσει να κατέχει ακόμα τη δυνατότητα χρήσης του λιμανιού στο Κίεβο δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να την αγκαλιάσουμε. Θα πρέπει μάλλον να πούμε ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε να λέει ο Πρωθυπουργό ο κ. Λάμπροφ ότι δεν είναι προ τη τη Ρωσία να ενταχθεί η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίμιση των Ουκρανών υποστηρίζουν στερότερε σχέσει τη ε, χώρα του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να μην ανταποκριθούμε θετικά στι προσδοκίε του. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, εγώ σα ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στα πλαίσια των διακοινοβουλευτικών συνεδριάσεων μας έχουμε μία αντιπροσωπεία από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.